Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται διότι υπερβαίνει την πλειοψηφία των τριών πέμπτων των ψηφισάντων. Προχωρούμε στην επόμενη έκθεση, έκθεση ΚΟΧ με θέμα... Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Uh, Δεν λειτουργεί το μηχάνημά μου. Ένα τεχνικό ήθελα, παρακαλώ. Τεχνικός, μάλιστα. Προχωρούμε στην έκθεση ΚΟΧ ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφοφορία μονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προχωρούμε στην έκθεση Μιχαήλοβα, εδαφικές τυπολογίες από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τροπολογία 1, ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η πρώτη ανάγνωση ολοκληρώθηκε. Έκθεση Μέισνερ με θέμα αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοεία Τροπολογία 131. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η πρώτη ανάγνωση. Ολοκληρώθηκε. Έκθεση Σενάλοβα με θέμα συνεργασία παρακαλώ. Να διαβάσω τον τίτλο. Θα σας δώσω το λόγο με θέμα συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Το λόγο έχει ζητήσει η κυρία Ρέντα εκ μέρους της ομάδας των Πρασίνων. Κυρία Ρέντα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θέλω να προτείνω να ψηφίσουμε τις τροπολογίες πρώτα στο νομοθετικό κείμενο και μετά να δώσουμε την ευκαιρία στους ευρωβουλευτές να εντάξουν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα λοιπά Την ισχυρή αυτή θέση για την προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Την πρόταση της κυρίας Ρέντα θα ήθελε το λόγο επ' αυτού η συγγήτρια. Δεν ζητά το λόγο, επομένως... Α, παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Συνάλογα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι κατά της πρότασης ως εισηγήτρια. Προτείνω να ψηφίσουμε την τελική συμφωνία που απορρέει από τις νομιλίες. Σε ψηφοφορία την πρόταση της κυρίας Ρέντα όπως την ακούσατε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται να κάνουμε τσέκ αφού ζητήθηκε αν και ήταν καθαρή η απόσταση υπέρ αρχίζει η ψηφοφορία λήξη ψηφοφορίας η πρόταση απορρίφθηκε προτείνω να προχωρήσουμε επομένως αμέσως στην ψηφοφορία επί της τροπολογίας 151 με ονομαστική κλίση αρχίζει η ψηφοφορία λήξη ψηφοφορίας εγκρίνεται και η πρώτη ανάγνωση ολοκληρώνεται. Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Γκαρσία Πέρες «Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής αναπεριφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών». Η κυρία Γκαρσία Πέρες έχει δει το λόγο. Της δίνω το λόγο σύντομα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η Ευρώπη γερνάει. 80% του πληθυσμού είναι στο 20% της επικράτειάς μας. Η Ήπεθρος υποφέρει αγωνιά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτή η απερίμωση. Σήμερα λοιπόν θέλω εδώ στο σώμα να ζητήσω προσοχή στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος και χτες σε σχέση με το ζήτημα αυτό, όπου έλεγε ότι υπεύθυνοι της απερίμωσης αυτής είμαστε οι γυναίκες ότι εμείς φταίμε που πήγαμε να δουλέψουμε και δεν μείναμε στα σπίτια μας να κάνουμε παιδιά. Αυτό αποτελεί προσβολή κατά των γυναικών, οι οποίες είναι ελεύθερες. Είναι προσβολή απέναντι στις γυναίκες λοιπόν που είναι ελεύθερες να δουλέψουν ή να μείνουν στο σπίτι τους που είναι ελεύθερες να αποφασίσουν αν θέλουν να γίνουν μητέρες ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μελετήσει τις δηλώσεις αυτές για να δει κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρξει κύρωση σε βάρος ε, του κύριου Μίκε. Θέλω να σας πω επίσης ότι αυτός που θα έπρεπε να κάτσει σπίτι του είναι όλοι όσοι μισούν τις γυναίκες, που δεν τις σέβονται, εκείνες τις γυναίκες που, που είναι όπως όλοι, όλες εμείς που αποφασίσαμε να είμαστε ελεύθερες. Ο κύριος Γκόλνης έχει ζητήσει το λόγο επί Κύριε Γκόλνης, σας ακούμε. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το διαδικαστικό μου βασίζεται στο άνθρωπο που αναφέρεται στις κυρώσεις σε βάρος των Ευρωβουλευτών. Ε, να ξέρετε ότι δεν συμφωνώ πάντα με αυτά που λέει ο κύριος Κόρβιν Μίκε. Όμω, μια που πρόκειται για έναν παλιό Ευρωβουλευτή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν σα κρύβω ότι ανησυχώ με την τροπή, την κατασταλτική που έχουν πάρει τα πράγματα εδώ και που εμφανίζεται όλο και περισσότερο. Άλλοτε το Προεδρείο και ο Πρόεδρος μπορούσαν να επιβάλλουν κυρώσεις μόνο σε όσους εμπόδιζαν τη λειτουργία της Ολομέλειας. Τώρα όλο και περισσότερο φαίνεται ότι όποιος λέει κάτι που δεν αρέσει μπορεί να αποτελέσει θύμα κυρώσεων. Ποιος αποφασίζει αν αυτό που λέει είναι καλό ή κακό. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε μια τέτοια τροπή των πραγμάτων που είναι πάρα πολύ σοβαρή όπως και αυτή που έχουμε με το ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του κύριου Μπουτζεμόντ. Εγώ μπορεί να μην είμαι υπέρ τη ανεξαρτησία της Καταλωνία προσωπικά, αλλά δεν θεωρώ φυσιολογικό αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα να χρησιμοποιείται σε βάρο κάποιου πρόσφυγα, σαφώς πολιτικού πρόσφυγα. Κυρία Γκαρσία Πέρες, ως Προεδρεύων δεσμεύομαι να μεταφέρω και στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και στο Προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου την πρότασή σας να μελετήσουμε τις δηλώσεις του συναδέρφου Κόρβιν Μίκε και δεσμεύομαι να το κάνω και για έναν πρόσθετο λόγο ότι ανάμεσα στις αρμοδιότητες που έχω ως Αντιπρόεδρος είναι η προάσπιση της ισότητας των φίλων και νιώθω διπλή υποχρέωση να κάνω αυτό που προτείνατε. Προχωρούμε Α, ο κύριος Κόρβιν Μίκε θέλει το λόγο και πάλι. Μάλιστα κύριε Κόρβιν Μίκε. Ε, ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κυρία Γκαρισία Μπέρες έκανε κάτι το σκανδαλώδες αυτή τη στιγμή γιατί τάσσεται κατά της ελευθερίας της σκέψης που αποτελεί πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Προεδρείο νομίζω πως θα πρέπει να τοποθετηθεί από αυτό. Σας ευχαριστώ. Για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική κλίση αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προχωρούμε στην έκθεση Λούντβιξον σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για το σύνολο του κειμένου ψηφοφορία με ονομαστική κλίση αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Προχωρούμε στη διαδικασία αιτιολόγησης ψήφου. Α.